Okay, Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλημέρα σας. Ας εγκρίνουμε καταρχάς την ημερήσια διάταξη, την οποία την έχετε στους φακέλους σας. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία, εγκρίνεται. Δεν προβλέπονται ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο. Συνεπώς, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 6ης και 7ης Μαΐου 2015. Και τα πρακτικά τα έχετε στο φακελό σας. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, ενημερώστε τη γραμματεία πριν το τέλος συνεδρίασης. Αν δεν λάβουμε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4. Έγκριση αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών. Έχετε λάβει πάλι το σχέδιο των συμπερασμάτων και των, συστάσεων των συντονιστών της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου. Αν έχετε παρατηρήσεις, ενημερώστε πάλι τη γραμματεία μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αν δεν λάβουμε και πάλι παρατηρήσεις, θα εγκρίνουμε τις αποφάσεις και τις συστάσεις των συντονιστών. Σημείο 5. Ανακοινώσεις της Επιτροπής. Υπάρχουν παρατηρήσεις από την Επιτροπή. Όχι. Επομένως κλείνει και αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης. Και περνάμε στο σημείο 6. Η κρίση του ιού του έμπολα διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό σημείο που πρέπει να εξετάσουμε στη μερίσια διάταξη. Θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την έκθεση του κυρίου Γκέρενς όσον αφορά την κρίση του ιού έμπολα. 157 συνολικά είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα πρέπει να ψηφίσουμε επίσης και τις ε, γνωμοδοτήσεις που έχουμε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Γκέρενς προκειμένου να μας παρουσιάσει τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την έκθεσή του. Τσάρλς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν ολοκληρώνουμε λοιπόν την εργασία μας για την έκθεση αυτή. Δεν μένει παρά να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες και να συμφωνήσουμε για τον, τη μέθοδο την οποία θα ακολουθήσουμε προκειμένου να ψηφίσουμε στη συνέχεια την έκθεση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ελπίζω ότι θα είμαι σε θέση να υποβάλω συμβαστικές τροπολογίες στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην επόμενη δηλαδή συνεδρίασή μας, και ελπίζω θα καταφέρουμε να εντάξουμε κάποια ολομέλεια και την έκθεση αυτή. Στόχος της έκθεσής μου ήταν να δούμε από κοινού πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη, την εξέλιξη του ιού του έμπολα, της νόσου αυτής και είχαμε συμφωνήσει όλοι στα πλαίσια της έκθεσης ότι η επέκταση του ιού αυτού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική Ουδέποτε είχαμε δει μια τέτοια επέκταση της νόσου σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ή να έχουμε τόσο μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Δεκάδες χιλιάδες άτομα έχουν εμολυνθεί από τον ιό αυτό με τις πολύ δεινές επιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν φυγεί από τον ιό αυτό. Αναφερθήκαμε επίσης πιο συγκεκριμένα σε τρεις χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται σε μια συγκρίσιμη οικονομική κατάσταση, κατάσταση όσον αφορά την ε, ευημερία των ανθρώπων, ξεπερνά το 80% η ε, ακραία φτώχεια στις χώρες αυτές, η φίτηση στα σχολεία στις τρεις αυτές χώρες είναι κάτω από τα τέσσερα χρόνια, ενώ το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται ανάμεσα στα 50 και 60 χρόνια. Είχαμε λοιπόν την ε, δυνατότητα να δούμε καταρχάς πώς αντέδρασαν οι χώρες αυτές, τι έγινε επί τόπου και τι έγινε σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Καταρχάς, δέχτηκε επικρίσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν του επικρίναμε όμως το γεγονός ότι ανέλαβε δράση γρήγορα στην αρχή. Ήταν από τον Σεπτέμβριο και μετά που τα πράγματα εξελίχθηκαν πιο γρήγορα και πιο άσχημα και ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο του 2014 εγκρίναμε ένα ψήφισμα, τότε κινητοποιήθηκε περισσότερο ο οργανισμός αυτός και προσπαθήσαμε επίσης να δούμε και τι έκανε προληπτικά η διεθνής κοινότητα προκειμένου στο μέλλον να αποφευχθούν τέτοιες κρίσεις από την εξέλιξη της κρίσης αυτής του ιού του έμπολα στις τρεις αυτές χώρες συνειδητοποίησαμε ότι ήταν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθούμε να δίνουμε τουλάχιστον 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τον τομέα αυτό της ε, υγείας, για τον τομέα της ανάπτυξης των συστημάτων υγείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι θύνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δούνε τι δυνατότητα τους δίνουν προκειμένου να επαναπρογραμματίσουν την χρηματοδοτική βοήθεια για τις τρεις αυτές χώρες, γιατί πραγματικά ο νόσος του έμπολα έχει ε, επιδεινώσει πάρα πολύ την κατάσταση στις χώρες αυτές. Έτσι λοιπόν από το 2014 και μετά τα όσα γνωρίζουμε για την εξέλιξη της νόσου αυτής δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην πρώτερη περίοδο όταν δηλαδή προγραμματίζαμε την ανθρωπιστική βοήθεια για τις χώρες αυτές, στα πλαίσια δηλαδή του ετήσιου ή πολιετού προγραμματισμού. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, στο μελλοντικό της δηλαδή προγραμματισμό, να λάβει υπόψη στη διάσταση αυτή, της ανάπτυξης δηλαδή των συστημάτων υγείας σε αυτές τις χώρες και είπαμε ότι θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει μια ομαδοποίηση των προσπαθειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και κυρίως σε ενωσιακό επίπεδο και ακριβώς Γι' αυτό το λόγο διορίσαμε τον κύριο Στυλιανίδη, επίτροπο αρμόδιο για την ανθρωπιστική ε, δράση και ο οποίος είναι και υπεύθυνο για το συντονισμό της δράσης αυτής καταπολέμησης του, της νόσου του έμπολα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν να τον βλέπουμε συχνά τον κύριο Στυλιανίδη προκειμένου να ενημερωνόμαστε από αυτόν για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και τέλος υπάρχει και το ζήτημα της αποκατάστασης, της ανοικοδόμησης της οικονομικής των τριών αυτών χωρών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την νόσο του έμπολα και που γνωρίζουν βέβαια και πάρα πολλές οικονομικές δυσχέρειες. Σε πολλές περιπτώσεις η οικονομία έχει παραλύσει εντελώς, προκειμένου λοιπόν να προκύψει μια οικονομική ανάκαμψη, προκειμένου να δημιουργηθούν εκ νέου επαρκείς πόροι στις χώρες αυτές, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το δημόσιο σύστημα, το σύστημα των δημοσίων υπηρεσιών, απαιτείται χρόνος και απαιτούνται και, χρήματα όμως. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει και μία διεθνής διάσκεψη δωρητών για την οικονομική ανάκαμψη των τριών αυτών χωρών. Όλα αυτά αποτελέσαν λοιπόν αντικείμενο συζήτησης και υπήρξε μια γενικότερη συνένεση μεταξύ ημών για όλα αυτά τα σημεία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν είδα ότι είχαν υποβληθεί τόσες πολλές τροπολογίες για την έκθεσή μου. Βέβαια, όταν υποβάλλονται πολλέ τροπολογίε, αυτό σημαίνει ότι περισσότερο περισσότεροι έχετε διαβάσει επισταμένο την έκθεση. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μελετήσατε την έκθεση αυτή. Βλέπω επίση ότι έχετε θέσει κάποια κέρια επιχειρήματα στα πλαίσια των τροπολογιών σας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και εγώ να επαναθεωρήσω κάπως τη στάση μου σε κάποια σημεία. Αναλάβατε ιδιαίτερα δραστήρια δράση, αναφέρομαι για παράδειγμα στον κύριο Μωρής Πόγκα, Ποιο θα το περίμενε, αλλά ο κύριο Πόγκα έδειξε ένα εξαιρετικό ζήλο. Ο Μωρή ε, τόνισε το ζήτημα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και επίσης ε, αναφέρεται στην ε, αναθεώρηση, στη μεταρρύθμιση που προβλέπεται στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2015, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά όλη την απαραίτητη κατάρτιση τα μέλη του ιατρικού προσωπικού και σε ορισμένε περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια να αμβληθεί λίγο η ευθύνη που φέρει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε τον οργανισμό αυτό. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καταπολέμηση πολλών και διαφόρων νόσων. Θα πρέπει να καταφέρω λοιπόν στα πλαίσια των συμβαστικών μου τροπολογιών να εντάξω κάπως και αυτές τις τροπολογίες του κυρίου Πόγκα. Επίσης ε, αναφέρεστε στο 11ο Φόρουμ Ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει και αυτόν το λάβουμε υπόψη μας προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα της ε, ανάκαμψης των συστημάτων ε, υγείας και πρέπει όμως να δούμε πώς θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει και να προσαρμόσει την δική της συμβολή. Αυτό το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι μια κάποια μαγική λύση, είναι μια ένδειξη, ενδεχομένως να μην φτάνει το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά οι τρεις αυτές χώρες που έχουν ε, πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του ιού έμπολα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε κάποιες βασικές κοινωνικές υπηρεσίες στις χώρες αυτές. Ο συνάδελφος κύριος Νόιζερ και αυτός υπέβαλε πολλές τροπολογίες. Λυπάται που στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης αναφερόμαστε μόνο στην Γουινέα, αλλά όχι στη Σιέρα Λεόνε και όχι στη Λιβερία, όσον αφορά δηλαδή την ανάπτυξη των υγειονομικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν έχει δίκιο ο κύριος Νόιζερ, ότι δηλαδή έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη Γουινέα μόνο και όχι στις υπόλοιπες ε, χώρες. Από τους Πρασίνους η κυρία Σαρτζετίνη και Ριβάζη αναφέρονται στις δεινές συνέπειες που είχαν ε, τα προγράμματα αποκατάστασης ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης παιδείας και ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον κλάδο αυτό στις τρεις αυτές χώρες. Πραγματικά Έχετε δίκιο. Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε στα πλαίσια της έκθεσης να συμπεριλάβουμε και τις παρατηρήσεις αυτές. Νομίζω ότι υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί παράγοντες που εξηγούν την κατάσταση και το γεγονός ότι δεν έχουν συμβάλει αρκετά, δεν έχει συμβάλει αρκετά η διεθνής κοινότητα όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί αν είχαν δοθεί τα παρέτα κονδύλια επαρκώς από τη διεθνή κοινότητα θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις ε, καταστροφικές συνέπειες τις δράσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πάντως συνάδουν οι δικές σας τροπολογίες όσα λέω και εγώ στην έκθεση. Ο Λί Μισελ στη συνέχεια αναφέρεται στο, στην ομαδοποίηση κάπως των κρίσεων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δεκτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε αυτές τις χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα από τις τροπολογίες αυτές ενισχύεται τα βασικά σημεία, τις βασικές προτάσεις που γίνονται στην έκθεση αυτή. Είναι όντως πολλές τροπολογίες, χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό και στα πλαίσια ενός επικοδομητικού πνεύματος θα ήθελα να συντάξω στο μέλλον κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Έχω ήδη κάποιες πρώτες ιδέες, αλλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου τις συμβαστικές με αυτές προτάσεις ε, στα πλαίσια μιας επιτροπής μικρότερης έτσι σύνθεσης. αλλά θα μπορούσαμε ακόμα και τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε ένα πιο σύντομο κείμενο συμβαστικών τροπολογιών. Αυτές είναι οι αρχικές μου αντιδράσεις όσον αφορά τις τροπολογίες που καταθέστηκε για την έκθεσή μου και προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες παρατηρήσεις. Σε ευχαριστώ Σάρλ. Να ακούσουμε τώρα τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Πόγκαθ είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάγλ. Θα ήθελα να ανατετυπώσω τα σημεία που ανέφερες σε σχέση με τις δικές μου τροπολογίες στην έκθεσή σου. Καταρχάς, να σε συγχαρώ για την δουλειά που έκανες για τον νέο του έμπολα. Νομίζω 27 τροπολογίες έχω καταθέσει. Όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση για τις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσα. Κατέθεσα λοιπόν τροπολογίες για να διευκρινίσω ορισμένα σημεία και να θυμίσω τη συμμετοχή της Ένωσης και ιδίως του Επιτρόπου κ. Στυλιανίδη και τη δράση του στο πλαίσιο της κρίσης, όπως και εσύ υπογράμμισες. Επίσης ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιφυλακής απαγρύπνησης ε, στην, ε, για να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά και στο μέλλον με τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων. Έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε υγειονομικές ε, τέτοιες καταστάσεις και να μπορούμε να τα αποκριθούμε τάχιστα, κάτι το οποίο δεν έγινε το Μάρτιο με τον ιό του έμπολα. Ένα άλλο σημείο που και εσύ υπογράμμισες και θεωρώ και εγώ σημαντικό είναι το ζήτημα της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ ε, των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μοιραστεί την εμπειρία της, τις επιστημονικές ιατρικές της γνώσεις. Πρέπει να διανεμηθούν, να διαβιβαστούν και στο ιατρικό προσωπικό των χωρών αυτών για να αποφύγουμε μια νέα πανδημία και σε ό,τι αφορά το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, ένα μέρος του θα πρέπει να πηγαίνει σε επενδύσεις ε, στον ιατρικό τομέα. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι ορισμένες από τις παρατηρήσεις μου, αλλά επαναλαμβάνω έχει την πλήρη υποστήριξή μου, μπορεί να βασίζεσαι σε μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής ε, είναι ο κύριος Νόιερ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Τσάρλς ε, για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Ε, εμείς βεβαίως ε, καλή έκθεση περιμέναμε από σένα. Ανέφερες πολλές τροπολογίες και νομίζω αυτό οφείλεται στο ότι όσον αφορά το θέμα αυτό ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ όλα τα μέλη. Νομίζω ότι η έκθεση αγγίζει τις ρίζες ε, του προβλήματος ε, και κατ' ουσίαν έχει και μια ενεργό προσέγγιση για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους επιδημιών. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση ε, παραμένει επίκαιρη και εδώ και κάποιες ημέρες πολλοί αναφέρουν ότι έχουμε και πάλι 30 νέα κρούσματα του έμπολα. Όμως ε, οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν είναι αυτοί που είχαν ήδη μολυνθεί, είναι άγνωστο από πού προήλθαν αυτά τα κρούσματα. Άρα δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με τον έλεγχο. Και νομίζω ότι από τις τροπολογίες προκύπτει ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας ε, σε αυτές τις χώρες και πρέπει να διαθέσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Η αναπτυξιακή βοήθεια, εκεί πρέπει, αυτό πρέπει να είναι σαφές, ότι οφείλουμε ε, την αναπτυξιακή βοήθεια να τη δίνουμε για ε, υποδομή, για έργα υποδομής. Αν δεν υπάρχουν αν δεν υπάρχει πρόοδος ε, σε αυτόν τον τομέα, εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε παρόλα αυτά σε αυτό. Και κατά τα άλλα πιστεύω, πρέπει να αναφέρουμε ότι στις χώρες εταίρους θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη περίθαλψη υγείας. τα κονδύλια να δαπανώνται και για την ε, περίθαλψη υγείας. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διάλογος. Πριν από ε, τέσσερις περίπου εβδομάδες ε, είχαμε την G7 στη Γερμανία. Ετέθη το θέμα και αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει η αντιμετώπιση υγείας μέσα από ένα κρίκο που αφορά και τον άνθρωπο και τα ζώα σε αυτή την συνάντηση κορυφής ε, G7 ε, και δεν πρέπει να το κρύβουμε. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, για μένα τουλάχιστον, ήταν στραμμένες οι αποφάσεις ε, περισσότερο προς τον αξιονισμό, όπως το να προκαλέσουν εντύπωση και δεν ήταν επί της ουσίας οι αντιδράσεις ήταν όπως αυτές που διαπιστώνει κανείς στο στρατό. Δηλαδή κάτι έγινε, κάτι πρέπει να κάνουμε και θα τα ελέγξουμε όλα. Δηλαδή με λίγα λόγια καμία ε, μελλοντική προσέγγιση. Δεν υπήρχε το στοιχείο της διάρκειας σε αυτές τις αποφάσεις των G7. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις αποφάσεις της, της ε, Κομισιόν του 2010 ε, εκεί προβλέπεται ενίσχυση των ε, συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο και επίσης προβλέπεται να υπάρχουν και ουσιαστικά αιτήματα σε αυτή την ατζέντα για θέματα υγείας που προτιθέμεθα να θέσουμε επιτάπητος. Το θέμα λοιπόν το οποίο αφορά την, ε, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ετέθη και πιστεύω ότι στο μέλλον ο ΠΟΗ ε, θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι κυρίως όσον αφορά την βασική έρευνα, οφείλουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτήν. Χρειαζόμαστε νέες δραστικές ουσίες, γιατί η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι ένα πρόβλημα και αυτό ετέθη επίσης στην ε, διάσκεψη των G7. Άρα δηλαδή περισσότερα κονδύλια για να ε, προωθηθεί η βασική έρευνα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Επίτροπός μας για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, ο κύριος Τηλιανίδης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε μαζί του το συνεχή διάλογο για να παραμείνει το θέμα επίκαιρο. Άρα δηλαδή η Επιτροπή μας οφείλει να φέρει και να επαναφέρει το θέμα ε, να το συζητάει με τον Επίτροπό μας, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά στο θέμα της αντιμετώπισης του έμπολα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Σάρλ για την έκθεσή του. Ο Νόρμπερτ Νόισερ πολύ σωστά είπε ότι παραμένει επίκαιρο το θέμα. Νομίζαμε ότι η Λιβερία έχει απαλλαγεί πλέον από τον ιό του έμπολα, αλλά δεν σημαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει, αυτό. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να ε, εργαζόμαστε για την ανικαδόμηση αλλά να μην καθυστερήσουμε. Και ίσως δεν είναι και το μόνο πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δούμε. Έχουμε τη φτώχεια, έχουμε τις ασθένειες αυτές ε, και την κακή διαχείριση και την κακή οικονομική κατάσταση. Καταστροφή είναι το αποτέλεσμα και έχουμε ε, ένα τέτοιο παράδειγμα αυτές τις χώρες. Και η Παγκοσμία Οργάνωση Υγείας δεν φαίνεται να κάνει αυτά που ε, πρέπει. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και ακόμη χειρότερα. Και Χάρη στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις κυρίως ε, δεν ήταν ακόμα μεγαλύτερη κρίση. πράσινη στις τροπολογίες μας έχουμε εστιάσει στην ε, αναδιάρθρωση και στην επιρροή των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Διότι για μας αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η χώρα, μια χώρα δεν μπορεί να είναι ανθεκτική όταν γίνονται περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα υγείας. Τότε ο πληθυσμός, η κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κρίσεις. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό να το δούμε αυτό το θέμα σε ένα ευρύτερο πακέτο, σε μια ευρύτερη δέσμη προτάσεων, διότι αλλιώ είτε με την ίδια νόσο ή με ε, μια διαφορετική μεταδοτική νόσο θα δούμε ξανά τα ίδια. Αν μπορούμε λοιπόν να, να εργαστούμε από κοινού με τον ΣΑΡ για συμβαστικές τροπολογίες ε, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Γιατί έτσι θα έχουμε μια ευρύτερη εικόνα της δράσης μας. Επίσης, και στην ετολική σου έκθεση, Σαρλ, και στην έκθεση αναφέρεσαι στην κρίση μέσα στην κρίση. Δηλαδή, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναστούν βοήθεια για μια άλλη νόσο. Και έτσι δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αντιμετωπίζονται άλλα προβλήματα υγείας. Οπότε η κοινωνία πάσχει ακόμη περισσότερο και γίνεται λιγότερο ανθεκτική και στην αντιμετώπιση κρίση και στις ασθένειες. Η έκθεση και οι τροπολογίες Γιατί όπως είπε και ο Νόρμπερτ, ε, οι τροπολογίες δείχνουν ότι ενδιαφερόμαστε για την έκθεση, είχαμε ενδιαφέρον για την έκθεση. Η Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να δει όμως ε, ευρύτερα, με ευρύτερη προοπτική και όχι με στενή προοπτική να δούμε ποια ήταν τα γεγονότα και να τελειώνουμε. Όχι. Ε, μας ενδιαφέρει και η ανοικοδόμηση τριών χωρών από πολύ δύσκολες συνθήκες και σε ένα δύσκολο περιβάλλον στη Δυτική Αφρική. Μετά το καλοκαίρι θα τα ξαναπούμε. Ευχαρίστω Thank you. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάποιο ε, συνάδελφο από κάποια ομάδα, αλλά θα ήθελα να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να απαντήσετε, ενδεχομένως να κάνετε κάποια σχόλια μετά από τη συζήτηση που ακούσατε, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουμε γρήγορα σε σχέση με την έκθεση. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει, ε, είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην αντιμετώπιση του έμπολα με διάφορες γενικές διευθύνσεις. Και είναι πρόσδεκτο το σώμα της έκθεσης, ε, γιατί πιστεύουμε ότι ασχολείται με τα βασικά σημεία, τα καλύπτει και θεωρούμε ότι σε πολλά σημεία της εκθεσής σας υποστηρίζεται και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά μέσα από τι ανησυχίε που εγείρεται στην έκθεση, νομίζω ότι εν μέρη αντιμετωπίζονται για την ε, διάσκεψη των ε, χρηματοδοτών έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. 450 εκατομμύρια προτείναμε για τις τρεις πληγήσεις χώρες και την ανοικοδόμησή τους. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα Επανεξέταση ε, θεώρησης του προγράμματος για τις τρεις αυτές χώρες, οι αντιπροσωπείες μας και οι υπηρεσίες μας είχαν ε, επαφές ε, με τις εθνικές αρχές στις τρεις αυτές χώρες. Οι αρχές όμως των ελόγων χωρών μας ξεκαθάρισαν ότι έχουμε αυτούς τους δημόσιους τους κανονισμούς Έχουμε και άλλους εταίρους που μας υποστηρίζουν ιδίω στον τομέα τη υγεία ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υποστηρίζει σε άλλου τομεί. Άρα είναι συμπληρωματική η βοήθεια. Οι εθνικέ αρχέ, λοιπόν για αυτό το κύκλο προγραμματισμού 2014-2018 δεν υπέβαλαν έτοιμα για ε, να ξανανοίξουμε τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα. Έχουμε τον εστιακό μας ε, τομέα για την υγεία στη Γουινέα γιατί η Λιβερία και τη Σιαρελόνε δεν έχει γίνει υγεία ε, στιακός τομέας. Και για τη Σιέρα έχουν και τη μακροοικονομική βοήθεια, μεταφορές, ασφάλεια τροφίμων. Ε, εστιάζουμε σε κοινωνικούς τομείς ε, στις τρεις αυτές χώρες ε, αλλά στον τομέα της υγείας και της παιδείας γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δραστηριοποιούνται στη Λιβερία, ιδιαίτερα και το Ηνωμένο Βασίλειο στη Σιέρα Λεόνε για τον τομέα της υγείας και έχουμε αυτή την πολιτική επιμερισμού των βαρών ε, και εστίαση συγκεκριμένου τομεί. Άρα το πρόγραμμά μας ε, προς το παρόν παραμένει ευθυγραμμισμένο με τους στόχους αυτούς. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις ε, ε, χρηστής διακυβέρνησης, ε, βλέπουμε όρους που αφορούν την υγεία και που σχετίζονται με την εκταμείευση της διονομικής υποστήριξης. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας προς το παρόν τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Προτινόμενες τροπολογίες νομίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό ε, αντικαθρεπτίζουν τις ε, απόψεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τροπολογία 51 ε, τώρα μιλά για προθυμία των κρατών μελών και ανεπαρκή συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι τα πράγματα. Σίγουρα μπορεί να σκεφτεί κριτική σε όλους για την καθυστερημένη ανταπόκριση και αντίδραση στις πρώτες φάσεις της επιδημίας. Η ΓΑΜΑ ΕΚΟ όμως αντέδρασε πολύ έγκαιρα. Ε, είχαμε συντονισμό των γενικών διευθύνσεων. Νομίζω ότι και στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΟ που κάναμε μια συνάντηση απολογισμού είδαμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό και από τα κράτη-μέλη που ενέκριναν σε πολύ μεγάλη, ε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία τον τρόπο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες όπως η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία της ευρωπαϊκή Ένωσης και τι ρόλο έχει σε ό,τι αφορά κάποιες ερευνητικές προτάσεις. Θα μπορούσαμε ε, να δώσουμε πληροφορίες για τη διόρθωση των πραγματικών περιστατικών. Μπορούμε να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες αν θέλετε όπως και για το θέμα των γυναικών και του έμπολα. Σίγουρα είναι σε θέση από πολλές οπτικές γωνίες οι γυναίκες ό,τι αφορά τον ιό του έμπολα και σε σχέση με τα στοιχεία που έχουμε δεν έχουμε ενδείξεις ότι πλήττονται περισσότερο γυναίκες είτε μεταξύ του γενικού πληθυσμού είτε μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Δεν θέλω όμως να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θελήσετε να σας υποβάλουμε περαιτέρω στοιχεία, τα οποία κρίνετε χρήσιμα. Ευχαριστώ. Εμείς... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι πήρανε όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην αίθουσα το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το γεγονός ότι υποβάλατε και διατυπώσατε τροπολογίες. Σε τέσσερα σημεία θα εμείνω. Όσον αφορά το ζήτημα της διαρθρωτικής προσαρμογής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν αλλάξει τη στάση τους από τη δεκαετία του 90 μάθαν από τα λάθη τους, προσαρμόσαν την πολιτική τους. Πρέπει να δούμε αν η νέα πολιτική είναι σωστή, αν επαρκεί, αλλά θα πρέπει και από την άλλη πλευρά και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε κάποια όρια, κάποια κατόφλια κάτω των οποίων δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στους πληθυσμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν μπορούμε να περιορίζουμε τα όσα προβλέπονται για τα δημόσια συστήματα υγείας. Τα συστήματα υγείας, η παροχή γενομικών υπηρεσιών αποτελεί ένα δικαίωμα ανεφέρετο το οποίο θα πρέπει να παρέχουμε με τη μορφή όλων αυτών των υπηρεσιών στους λαούς των χωρών αυτών. Υπάρχουν λοιπόν κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν πρέπει να ξεπεράσουμε. Και το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων και της πρόσβασης στα φάρμακα αυτά. Το ζήτημα της πρόσβασης των φαρμάκων μπορούμε να το επιλύσουμε πιο εύκολα και ήδη έχουμε σημειώσει πρόοδο στον τομέα αυτό στα πλαίσια της συμφωνίας TRIPS. Θα πρέπει όμως ε, να την παρακολουθούμε και την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Δεύτερον όμως τώρα, ποιος είναι ακριβώς υπεύθυνος για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων. Ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό στα πλαίσια της εταιρολογικής έκθεσης αλλά και στα πλαίσια του διατακτικού της έκθεσης αλλά και εσείς ασχοληθήκατε με το ζήτημα αυτό. Έχουμε προφανώς την φαρμακοβιομηχανία από τη μία πλευρά, η οποία αναπτύσσει φάρμακα με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται, επενδύει λοιπόν στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά από την άλλη έχουμε κάποιες νόσους οι οποίες δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο απαραίτητο εκείνο επίπεδο προκειμένου οι φαρμακοβιομηχανίες να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες και να αναπτύξουν νέα φάρμακα για αυτές τις ασθένειες, για αυτές τις νόσους. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το ζήτημα αυτό έχει να κάνει τόσο με τις επαγγελματίες του τομέα της υγείας, αλλά και με την πολιτική που ακολουθείται για τον τομέα αυτόν. Δεν έχω βαθύνει περισσότερο στην εκθεσή μου στο ζήτημα αυτό, πάντως νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή, καθώς επίσης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ιδιαίτερα πολύπλοκο και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε εκτενώς να το αναπτύξουμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να απτύξουμε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος αυτού στα πλαίσια της δικής μου της έκθεσης. Πάντως νομίζω ότι το ζήτημα αυτό της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων θα πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια μιας άλλης έκθεσης. Εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να σοπάσουμε πέντε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ο συνάδελφος Νόιζερ αναφέρθηκε στο G7. Όντως το G7 λειτουργεί πολύ αργά η πρόοδος πολλές φορές υστερεί πολλές φορές των πραγματικών επιθυμιών που έχουμε και βλέπουμε πολύ συχνά ότι το G7 μας σερβίρει ουσιαστικά κάποιες ε, αδύναμες, ε, δειλές πολιτικές. Σαφώς αυτό μπορούμε να το επικρίνουμε, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο πιο ενεργά με τις αποφάσεις που λαμβάνει το G7. Οι αποφάσει αυτέ είναι πολύ σημαντικέ, όχι μόνο για το τι πρόκειται να γίνει, αλλά για το τι δεν γίνεται πολλέ φορέ. Σε σχέση λοιπόν με τι αποφάσει που λαμβάνει το G7 θα πρέπει και εμεί να αντιδρούμε προκειμένου να ενημερώνουμε καταλήλω το G7 για αυτά τα οποία παραλείπει τελικά να κάνει. Ο κύριος Νόιζερ έρχεται από μια χώρα που διοργάνωσε πρόσφατα στην Βαβαρία το G7 και οι συναδελφοί σου από το Τσεντεού έχουν καλύτερες σχέσεις ενδεχομένως με την Καγκελάριο. Νομίζω ότι και εσείς αλλά και ο κύριος Πόγκα που προέρχεται από μια χώρα που συμμετέχει στο G7 αλλά και ο Βρετανός και ο Ιταλός συνάδελφος θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους πολιτικούς ηθήνοντες στις χώρες τους προκειμένου στα πλαίσια του G7 να καλύπτε περισσότερο το ζήτημα αυτό που μας απασχολεί σε αυτή την έκθεση. Όσον αφορά τώρα τη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών, θα πρέπει να ασχοληθούμε προφανώς και με το ζήτημα των γυναικών. Θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο τις γυναίκες στα πλαίσια τροπολογιών αυτών και να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο πολύ κέριος ρόλος που δραματίζουν ιδίω στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία των ε, νόσων αυτών και όσον αφορά το ζήτημα της ευαισθητοποίησης των παιδιών και του γενικού τροπληθισμού. Λοιπόν, απομένει να κάνουμε σημαντική ακόμα δουλειά στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Λυπάμαι πάντως, διότι από τη στιγμή που σταματήσαμε να έχουμε νέα κρούσματα έμπολα, σταματήσαμε να ασχολούμεθα πλέον με το ζήτημα του έμπολα στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και ότι θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα μετριοπαθείς και ταπεινοί απέναντι στο ζήτημα αυτό της κρίσης του ιού έμπολα. Όταν μιλήσω για την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια, θα θίξω και το εξή ζήτημα. Τι κάναμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχαμε 20.000 κρούσματα, 20.000 ανθρώπους οι οποίοι θα είχαν μολυνθεί από τον ιό έμπολα. Φανταστείτε να είχαμε τον αριθμό αυτών ανθρώπων που θα είχαν ασθενήσει από τον ιό τον έμπολα στις Βρυξέλλες. Τι θα κάναμε στην περίπτωση αυτή, πώς θα είχαμε αντιδράσει. Ας είμαστε λοιπόν αρκετά μετριοπαθείς και ταπεινόφρονες. Αναφερόμαστε πολλές φορές μόνο στα θύματα κάθε φορά που είμαι για την Αφρική. Ξεχνάμε όμως όλους αυτούς που ανέλαβαν ηρωική πραγματικά δράση, όλους αυτούς που με το κουράγιο τους, με το θάρρο τους κατάφεραν να σώσουν πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε κάθε φορά που μιλάμε για το ζήτημα αυτό. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερη ευχαρίστηση το γεγονό ότι κατάφερα να έχω μια γόνιμη συνεργασία μαζί σα. Από κοινού καταφέραμε να παραθέσουμε όλε αυτέ τις πολύτιμες ιδέες στα πλαίσια αυτή τη έκθεση, αλλά μην ξεχνάμε ότι φέρουμε και ότι θα φέρουμε και στο μέλλον μια πολύ σημαντική ευθύνη όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης της μετάδοσης του ιού του έμπολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα και πολύ πιο αποτελεσματικά μέτρα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, Τσάρλς. Θα συνεχίσουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις με τους και Τα Θα έχουμε ε, ψηφοφορία για αυτή την έκθεση 21-22 Σεπτεμβρίου. Και τώρα το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ο προϋπολογισμός. Όμως ο κύριος Φερνάντες ε, δεν είναι εδώ και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς εκείνο. Θα πρέπει να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Θα έρθει 11 παρα 25. Διάλειμμα για ένα τέταρτο. θα είναι εδώ 10 και 5. Άρα ε, διάλειμμα ένα τέταρτο.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 Okay.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 Θα συνεχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας, αλλά πριν περάσουμε στο ζήτημα του προπολογισμού, μία σύντομη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Νίλ δεν ήταν εδώ στην αρχή, μου ζήτησε να του δώσω το λόγο, παρακαλώ κύριε Νίλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας. Γνωρίζω ότι πολλοί βουλευτές της Επιτροπής σας, αλλά επιτροπής Επιτροπή σας, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την συνεκτικότητα της πολιτικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα για το σκέλος του εμπορίου. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μόλις ε, μία πολύ καλή έκθεση για την αξιολόγηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων των εμπορικών καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες, ανψόμενες χώρες. Αξιολόγηση οικονομικών λοιπόν ωφελών που προέρχονται από τα εμπορικά καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες επαναλαμβάνει τον τίτλο μιλητής. Είναι και περιγραφικός ο τίτλος. Είναι ενδιαφέρουσα καλογραμμένη έκθεση με μια μεθοδολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων και πολλών άλλων ε, εργαλείων της εμπορικής πολιτικής μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορεί να γνωρίζετε ότι το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγάλο είναι μια τεράστια αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες αυτές, 86 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Ιδίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που είναι ακόμα πιο μεγάλο αυτό μερίδιο. Αν θέλετε έχω και έντυπα αντίγραφα μαζί μου Αλλιώς μπορείτε να βρείτε την έκθεση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Ε, είναι φρέσκια έκθεση, την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε. Η ΓΑΜΑ ε, Trade, ΤΕΦΚΟ, ΤΑΞΟΥΤ, ε, τα Copenhagen Economics, Λουβά, το Πανεπιστήμιο της Λουβάν και άλλοι ακαδημαϊκοί ερευνητές έχουν συνεισφέρει. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πω. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίλ. Σας ευχαριστούμε και για την έκθεση που με τα χαρά θα την μελετήσουμε. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της μερικής διάταξης, στον προϋπολογισμό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο έτος. Και θέλουμε να προετοιμάσουμε τις ετροπολικές μας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να ε, διεξαγάγουμε τα λόγου γνώσεως ε, της ε, προσεχής μας συζητήσης. Το Συμβούλιο έκρινε τη θέση του την προηγούμενη εβδομάδα και ο συνήθως ε, προέβησε σημαντικές περικοπές σε σχέση με τις προτάσεις ε, της Κομισιόν. Ευτυχώς, όχι για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να μην γίνουν περικοπές, λαμβάνοντας υπόψη το, τη Συρία, την, τη, το Νότιο Σουδάν, την κατάσταση εκεί, Υπήρχε όμως, αν θυμάστε καλά, κενό πληρωμών και γινόταν μεταφορά εις νέων από χρονιά σε χρονιά. Εμείς έχουμε μαζί μας τον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες ε, που είναι ο γενικός ηγητής, ε, συνεισηγητής μάλλον για τον γενικό προπολογισμό. Θα μας μιλήσει περίπου 30 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και θα έχουμε αφού μιλήσει ο ίδιος την ανταλλαγή απόψεων. Αν είναι ο δικός μας εισηγητής, θα μιλήσει μετά για να μας πει την άποψη της δικής μας Επιτροπής και τη γραμμή που προτίθεται ίδιος να ακολουθήσει. Ο κ. Φερνάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω περάσει από όλες τις επιτροπές, η δική σας είναι η τελευταία στην οποία παρίσταμε. Και έχω έρθει εδώ για να ακούσω και τις δικές σας πληροφορίες, τα δικά σας στοιχεία, για να καταρτήσω τον καλύτερο δυνατό περιπολισμό με τη δική σας βοήθεια. Σήμερα ήδη έχουμε τριμερή διάλογο και με το Συμβούλιο για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σας επενθυμίζω ότι εγκρίναμε στην Ολομέλεια τα guidelines, τις κατευθυντήριες γραμμές, και στην ε, τελευταία ολομέλεια έλαβα εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι σαφείς οι προτεραιότητές μας. Τα τρία ή ε, απασχόληση επιχειρήσεις και δι μικρομεσαίες και επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό πνεύμα, εσωτερική αλληλεγγύη και εξωτερική αλληλεγγύη βέβαια είναι πολύ σημαντικές πτυχές. Δεν ε, πρέπει να ξεχνάμε την συμφωνία του, την σημασία του προπολογισμού και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το όσα συμβαίνουν στη Συρία, στο Σουδάν κτλ. Τέλο πάντων γύρω από την Ευρώπη και στον κόσμο ευρύτερα. Το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπευλήθη στις 27 Μαΐου. Το Συμβούλιο συνήθως προτείνει περικοπές. Ευτυχώς στον τομέα το δικό σας δεν ε, θίγονται παρά λίγα κονδύλια. Υπάρχουν όμως κάποιες περικοπές τις οποίες κρίνω απαράδεκτες. Είναι μικρός ο προπολογισμό μας, ε, γύρω στο 1% του ΑΕΠ. 20% του ΑΕΠ είναι στη ΣΥΠΑ ο προπολογισμό. Αλλά είναι σημαντικός ο προπολογισμό. 94% για επενδύσεις, 6% μόνο για διοικητικές δαπάνες. Προσθέμενη αξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού λοιπόν είναι τεράστια. Και αυτό μας δίνει ακόμη και αν είναι μικρός αυτός ο ε, μας δίνει τη θέση του πιο ε, σημαντικού χρηματοδότη ε, στον κόσμο σε πολλούς τομείς. Είναι κάτι που δεν το λέμε τόσο πολύ και δεν το γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας. Να σας αναφέρω επίσης το χρονοδιάγραμμα. 3 Σεπτεμβρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ε, από τους ε, εισηγητές 23 Ενάτου κατάθεση των τροπολογιών 28-29-30 ψηφίζουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών, 12-13 Οκτωβρίου ψηφίζουμε το ψήφισμα, 28 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Ολομέλεια και μέχρι τις 19 Νοεμβρίου υπάρχουν κάποιες εβδομάδες συνδιαλλαγής. Η αρχή είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις του το Συμβούλιο. Τι θα πει αυτό. Κοινοβούλιο και Επιτροπή έχουν καταλήξει συμφωνία σε ό,τι τα προβλήματα με τις πληρωμές. Και ελπίζω να την τηρήσει τη συμφωνία αυτή το Συμβούλιο, όπου σε αυτή τη συμφωνία το μέξο των ανεξόφλητων λογαριασμών για το 2016 είναι 2 δις. Το 2015 έχουμε 20 δις. Είναι ντροπή, όνειδος να μιλάμε για πληρωμές, πρόβλημα της πληρωμές ή δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα οι πληρωμές. Πάκτα sunt servanta. Ό,τι ε, το συμφωνούμε πρέπει να το τηρήσουμε. Είχαν συμφωνήσει και οι τρεις ε, και τα τρία θεσμικά όργανα για να υπάρξει λογαριασμός, τιμολόγιο, σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη κάτι. Άρα ε, πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για τέτοιο πρόβλημα. Και πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Δεν μπορεί να το συζητάμε συνέχεια στο Κοινοβουλίο αυτό το θέμα. Επίσης, αυτό το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο έχει εγκριθεί. Και έχουμε και την αρχή της ευελιξίας, τα μέσα ευελιξίας δηλαδή, που χρησιμοποιούνται. Ή ότι για πρώτη φορά είναι δυνατή η χρήση των περιθωρίων, δηλαδή μη ε, σε πιστώσεις των προηγούμενων ετών. Μέχρι τώρα δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή αναλήψη υποχρεώσεων. Ε, ό,τι περιθώριο δεν αξιοποιήθηκε εντάσσεται σε ένα γενικό ε, περιθώριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους βασικούς στόχους. Και κινούμε από αυτήν την αρχή ότι θα σεβαστεί το πολιτές πλαίσιο το Συμβούλιο και θα σεβαστεί και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Για να μην πω ότι θα έπρεπε να σέβεται τις ίδιες του τις διακηρύξεις και δηλώσεις. Γιατί είναι λογικό κάτι τέτοιο. Τώρα συγκεκριμένα. για τη δική σας την Επιτροπή. Στο σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύεται σημαντικά ε, τόσο η αναπτυξική συνεργασία και οι εθελοντικές ε, πρωτοβουλίες βοήθειας ένωσης και στις αναλήψεις υποχρώσεων και στις πληρωμές, το ίδιο ανθρωπιστική βοήθεια και το αποθεματικό για κατεπίγουσα βοήθεια. Στο αποθεματικό αυτό έχουμε αύξηση των πληρωμών. της τάξης του 106%. Βέβαια, εδώ έχουμε και το θέμα των ανεξόφυτων λογαριασμών, των απλήρωτων λογαριασμών. Στα κονδύλια που έχουμε περικοπές από το Συμβούλιο, εμείς ξεκινάμε από την καλή θέση και εγώ θα υπερασπιστώ τα κονδύλια και το σχέδιο προβλησμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Θα ήθελα να ξέρω και τις δικές σας προτεραιότητες. Να σας πω ότι στο μέσο συνεργασίας και ανάπτυξης 39,8 εκατομμύρια κόψη το Συμβούλιο 143 εκατομμύρια στις πληρωμές και για την πρωτοβουλία θελοντική βοήθεια εκεί 50.000 ευρώ μείωση. Συμβολική η δεν ξέρω γιατί το κάνει το Συμβούλιο. Είναι σαν να βάζει τα κονδύλια του προπολογισμού σε ένα μηχάνημα και υπάρχει κάποιες, ε, ε, στα κάποιες, Συντελεστέ στάθμισης και με κάποια κριτήρια κόβει από εδώ, από εκεί κτλ. Ε, όπως σας είπα, ανθρωπιστική βοήθεια και το αποθεματικό, το Emergency Aid Reserve, δεν έχουν υποστεί περικοπές. Φυσικά και πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους και για τα ε, κατεπήγοντα ε, ανθρωπιστικές κρίσεις. Μίλησα για την ευελιξία. Αυτά, αυτές είναι οι δικές μου θέσεις. Νομίζω ότι οι προτεραιότητές σας ε, εντάσσονται στην διαπραγματευτική μου εντολή. Δεν μπορούμε να λησμονούμε τη δική μας ευθύνη, πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σε ό,τι αφορά τους ε, εκτελεστικούς οργανισμούς, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν περικοπές 1% ε, το χρόνο. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά δεν μπορούν να υποχρεώσουμε τους εκτελεστικούς οργανισμούς. να εκπληρώνουν την αποστολή τους και αυτά που τους ζητάμε να τα φέρουν σε πέρας χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τους απαραίτητους πόρους. Πόσο κοστίζουν οι περικοπές, αυτό πρέπει να δούμε, γιατί περικοπές σε έναν οργανισμό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να φέρει σε πέρας κάτι και αυτό θα έχει κόστος και αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε αναοργανισμό, όχι οριζόντια. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερνάντες και τώρα θα ακούσουμε τις απόψεις της Επιτροπής. Έχουμε τέσσερα λεπτά για δύο μιλητές και ο πρώτος είναι ο κύριος Σφάτσενμπρούνα από την DG ECO. Ευχαριστώ κύριε... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που μόλις τώρα ακούσαμε από τον εισηγητή. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι πέρυσι είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά υπήρχε αυτή η ασφυξία στις πληρωμές, πολύ δύσκολα μέτρα ε, τα οποία ε, επηρέασαν ε, βέβαια κάποιες δράσεις που καθυστέρησαν και είχαμε και δυσκολία με τους εταίρους μας που δεν έλαβαν τα κονδύλια εγκαίρους. με τη δική σας βοήθεια πέρυσι μπορέσαμε κάπως να βελτιώσουμε την κατάσταση στον προϋπολογισμό. Και αυτή τη χρονιά υπήρχε ε, μια δικαιοσύνη, μια ισότητα στις πληρωμές ε, και τις ε, καταβολές. Μειώσαμε την προχρηματοδότηση για τους πιο ισχυρού εταίρους, κυρίως για τους διεθνείς οργανισμούς, τους αυτούς του ΟΗΕ και άλλους. Βέβαια, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να δίδεται σε πραγματικό χρόνο. Τα χρήματα χρειάζονται τώρα, εχθές δηλαδή, και αλλιώς δεν έχει νόημα η ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίξατε. Με τα μέτρα που προβλέπονται για φέτος ε, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το 15 έχοντας κατά νου την πρόταση της Επιτροπής ε, σχετικά με το να υπάρχει ε, πρικοδοτημένη γραμμή ανθρωπιστικής βοήθειας με περισσότερες πληρωμές από υποχρεώσεις κατ' ουσίαν ε, θα μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να απορροφήσουμε την καθυστέρηση πληρωμών που υπάρχει από την ε, προηγούμενη χρονιά ε, για λόγους που σας προανέφερα. Και μετά από αυτό θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση και θα μπορεί να χορηγείται η ανθρωπιστική βοήθεια λόγω κρίσης χωρίς ε, να υπάρχουν τεχνητές ε, καθυστερήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι η σημασία του γεγονότος ότι και το απόθεμα έκτακτης βοήθειας για την επόμενη χρονιά και αυτό έχει πρικοδοτηθεί επαρκώς. Αυτό δεν ίσχυσε φέτος ούτε και για παλαιότερα έτη. Μέχρι το 2012 αυτό δεν ήταν πραγματικό πρόβλημα, διότι κατά τη διάρκεια του έτους και σε διάφορες ε, πολιτικές είχαμε αρκετά υπόλοιπα πληρωμών τα οποία κατέστη δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ανθρωπιστική γραμμή, ε, στη γραμμή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, αυτό πέρυσι δεν ήταν δυνατόν διότι δεν υπήρχαν υπόλοιπα. Και οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή Προπολογισμού μας είπαν ότι ούτε και φέτος θα είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα υπόλοιπα. Και αυτό θα γίνει όπως σας είπα την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν για φέτος ε, και πάλι η βοήθεια έκτακτης ανάγκης ε, δεν ε, ισοδυναμεί πλήρως στα ποσά που υπάρχουν στις πληρωμές και τις υποχρώσεις. Δεν υπάρχει κάποια ρεαλιστική προοπτική έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνουν όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν η πρόταση είναι διαφορετική και έχουμε πλέον ε, πολύ καλή χρήση, δηλαδή ε, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε νέες καταστροφές, σε νέους σεισμούς, σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να μπορέσουμε και να ανταποκριθούμε και σε κρίσεις ε, που δεν προβλέπονται, αναφέρεται τις σημαντικότερες εξ αυτών. Επίσης, μετά την κρίση στη Συρία κατέστη απόλυτα σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νέες προτεραιότητες. Έχουμε 4 εκατομμύρια Σύριους που εγκατέλειψαν τη χώρα τους, 2,5 εκατομμύρια παιδιά και περισσότεροι εξ αυτών έχασαν τα πάντα. Έχασαν την πρόσβαση στα σχολεία και ως γνωρίζουμε αυτός είναι ο κίνδυνος σε μιας χαμένης γενιάς. Έχουμε ε, εντοπίσει νέες προτεραιότητες. Ο Επίτροπός μας ε, βρίσκεται σε επαφή μαζί σας και πρόσφατα ανακοίνωσε δημόσια ότι από τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς ε, το 3% του συνολικού προπολογισμού θα πρέπει να διοχετευτεί σε αυτές τις νέες προτεραιότητες. Και αυτό προστίθεται και σε όλους τους άλλους ε, περιορισμούς και σε ένα πολύ σφιχτό προπολογισμό που υπάρχει λόγω της ε, συνεχιζόμενης κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν με την υποστήριξη αυτής της καλής πρότασης της Επιτροπής και με το απόθεμα έκτακτης ανάγκης θα τα καταφέρουμε και ε, όπως είπατε και το Συμβούλιο το έχει ανακοινώσει αυτό. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα των τελικών διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2016. Και εμείς ευχαριστούμε από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ο κύριος Πάιχ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τα καθησυχαστικά του λόγια. Σε ό,τι αφορά την ΓΔ ΔΕΦΚΟ, ο προπολογισμό που καταθέσαμε είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προγραμματισμό που είχε γίνει. Αντικατοπτρίζει κάποιες ε, διακοιμάσεις, κάποιες παραλλαγές ε, σε σχέση με τις προτεραιότητες που είχαμε ορίσει. Είπατε ότι υπάρχουν ε, κάποιες συντελεστέ στάθμισης, κάποιοι αλγόριθμοι με τους οποίους με ένα μηχάνημα ορίζονται οι περικοπές. Όχι. Ε, εμείς ε, βλέπουμε τι διορθώσεις μπορούμε να κάνουμε από τη μια χρονιά στην άλλη και με βάση τις προτεραιότητες. Είχαμε τις προτεραιότητες μας στο πλαίσιο του πολιετούς προγραμματισμού και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Στη γραμμή ε, Νότια Αφρική, για παράδειγμα, προσπαθούμε να εστιάσουμε τη βοήθεια σε τέσσερα έτη μέχρι το 2017. Προσπαθούμε να έχουμε μπροστοβαρή ε, κατανομή ε, των κονδυλίων. Υπάρχει αυτή η βαθμιδόν προσέγγιση και στο τέλος καταργείται η συνεργασία. Εδώ έχουμε περικοπές πράγματι που σημαίνει ότι η πολιτική που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε δεν μπορεί να υλοποιηθεί αφενός και αφετέρου οι σχέσεις που είναι και αρκετά τεταμένες με την Νότια Αφρική ήδη ε, δεν θα βελτιωθούν και κατά ανάγκη. Λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με τη Λατινική Αμερική. Ε, εδώ έχουμε λιγότερες περικοπές μένα για τρεις χώρες όμως, Περού, η Σημερινό, Κολομβία. Ε, θέλαμε να, ε, τα συγκεντρώσουμε όλα, ε, γιατί και εκεί έχουμε αυτή τη βαθμιδόν προσέγγιση, όπου και εδώ τώρα βλέπουμε περικοπές. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι σημαντικές περικοπές ε, ε, στις αμοιβούς υποχρεώσεων είναι οι τοπικές αρχές. 13% περικοπές, 8 εκατομμύρια. Είναι ένα κονδύλιο που ήδη είχε πληγεί επειδή δεν είχαμε αρκετές πιστώσεις πληρωμών οι εταίροι πραγματικά αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα, πολλά έργα δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν ή χρειάστηκε να καθυστερήσει η υλοποίηση τους λόγω έλλειψης πόρων. Και εδώ πράγματι, αν, γίνει πράγματι αν γίνουν αυτές οι περικοπές, δεν θα μπορούμε να φέρουμε σε πέρα στην αποκεντρωμένη συνεργασία όπως είχε αποφασιστεί πολύ πρόσφατα. Τελευταία σημαντική περικοπή για τις δεσμεύσεις, αναλύσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων είναι το DCI. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν κάτω πάντα από το κατόφλι που προβλεπόταν. Τώρα, επειδή το DCI έχει μεγαλύτερη σημασία και αυξάνονται ε, τα, οι πληρωμές, ε, θέλαμε 5 εκατομμύρια παραπάνω που είχαν ε, κοπεί. Και τα χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά, γιατί υπάρχουν κάποια έργα που ξεκινάνε και θέλουμε να γίνουν διάφορες ε, μελέτες, ε, έλεγχοι και οτιδήποτε έχει να κάνει με την τρέχουσα διαχείριση των έργων αυτών. Τώρα έχουμε σπιστός πληρωμών. Δεν έχω την τύχη του συνάδελφου Βάλτερ δυστυχώς. Εδώ πράγματι στα κονδύλια Ντεύκο έχουμε μία τρύπα του 650 εκατομμύρια, 25% δηλαδή των πιστώσεων πληρωμών. Είμαστε στα μισά της χρονιάς και είμαστε ήδη στο 70% εκτέλεσης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την ασφάλεια των τροφίμων. Τη συγκεκριμένη γραμμή και άλλες έχουμε 90% φτάσει και θα έχουμε στο καλοκαίρι μέσα μάλλον ξεμείνει από χρήματα. για τον προϋπολογισμό τώρα της επόμενης χρονιάς. Ευθυγραμμίζεται με το κατόφλι του πολιτούς νοσονομικού πλαισίου και θέλαμε να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους καθυστερούμενους λογαριασμούς και τα τιμολόγια που θα έρθουν από εδώ και πέρα. Για να μην έχουμε την κρίση που έχουμε τώρα με τους ανεξαρτητούς και σίγουρα θα ξαναπροκύψει. Θέλαμε, είχαμε προβλέψει 600 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό είναι λίγο πολύ η τρύπα που θα έχουμε για φέτος. Το Συμβούλιο προτείνει και 200 εκατομμύρια περικοπές πάνω σε αυτά, άρα ευτυχώς θα έχουμε λιγότερα προβλήματα του χρόνου, όμως θα παραμείνει το πρόβλημα. Όπως και αυτή τη χρονιά είχαμε πρόβλημα και έχουμε πρόβλημα. Ε, πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και να έχουμε έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό. Και όπως είπε και ο κύριος εισηγητής, ε, με αυτό το προϋπολογισμό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να φέρουμε σε πέρα στις πολιτικές που έχουμε αποφασίσει. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you. Μάλιστα, εμείς σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Λίτς Ενδεχομένως όμως να πρέπει πρώτα να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν υποβάλουν ερωτήσεις στον κύριο Φερνάντες γιατί θα πρέπει να αποχωρήσει πριν το τέλος της συνεδρίασής μας. Έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις για τον κύριο Φερνάντες ή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια θα υπάρχει αρκετός χρόνος και αφού ακούσουμε και τον κύριο Λίτσε. Άουταλα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Φερνάντες, απευθύνομαι σε εσά. Μας είπατε ότι δεν ενημερώνουμε πάντα επαρκώς τους πολίτες για το γεγονός ότι ο σημαντικότερος χρηματοδότης παγκοσμίως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να ισχύει μεν, αλλά για παράδειγμα και η ίδια η Φιλανδία έχει μειώσει κατά 40% την δική της εθνική αναπτυξιακή βοήθεια και η κυβέρνηση της Δανίας πράττει αναλόγως. Αν λοιπόν αρχίζουμε τώρα να περηφανευόμαστε ότι είμαστε ο πιο σημαντικός δωρητής και χρηματοδότης παγκοσμίω, δεν θα ανταποκρίνεται πάρα πολύ αυτό στην πραγματικότητα. Μέσω αυτών των περικοπών τελικά διακυβεύεται και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι εταίρες μας. Μία εμπιστοσύνη την οποία με πολύ κόπο καταφέραμε να κερδίσουμε στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες θα είναι οι, περικο, περικοπές εξ ονόματος Συμβουλίου και ποιες είναι επιπτώσεις για τους εταίρους μας. Ο κύριος Νόιζερ έχει το λόγο. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες ε, και όπως το είπατε και εγώ πιστεύω ότι ε, πράγματι έχουμε μικρή πρόοδο ε, δηλαδή θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληρωμές που δεν έλαβαν χώρα εφόσον υπάρχει το εργαλείο της ευελιξίας. Δεν έχω να σας κάνω ερώτηση, απλά θέλω να σας πω τι ακριβώς γίνεται σε διάφορες αντιπροσωπείες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ε, υποσκάπτεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περικόπηκαν προγράμματα, καταργήθηκαν, αναβλήθηκαν και οι ΜΚΟ εκλήθησαν και μόνες τους να προκαταβάλουν κάποια ποσά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, με τον τρόπο αυτό, η αναπτυξιακή βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν επιθυμώ στην αντιπαράθεση με το Συμβούλιο να επισημάνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλές ε, αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εκφράζονται πολύ διπλωματικά, αλλά νομίζω ότι χάνεται η αξιοπιστία μας, γιατί κανείς πια ή πολλοί δεν μπορούν πια να μας υπολογίζουν λόγω αυτής της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, ασφυξίας εκ μέρους του ε, συμβουλίου. Ο κύριος Γκέρονς. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τις παρατηρήσεις του επίσημου συνεισηγητή μας, του κυρίου Φερνάντες. Πραγματικά χρησιμοποίησε τα καλύτερα λόγια για να περιγράψει την κατάσταση ως έχει. Όσον αφορά το προπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας καταρχάς, νομίζω ότι οι καθυστερούμενες πληρωμές μας δίνουν αρκετά στοιχεία αλλά δεν μας λένε πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα για την ε, χρηματοδότησή μας και για το πόσο τελικά αυτή είναι η κατάλληλη. Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές ε, καταφέρνουμε τελευταία στιγμή να εκταμιεύσουμε τα απαραίτητα κονδύλια όταν όμως προκύπτουν κάποιες έκτακτες ανάγκες για το 2014 και πολύ περισσότερο για το 2015 είχαμε δύο πολύ δύσκολα έτη. Ουδέποτε αντιμετωπίσαμε τόσες πολλές ανθρωπιστικές κρίσεις. Έχουμε τη Συρία, τη Λιβύη, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχουμε μία εκτίναξη των κρίσεων που πρέπει εμείς να καλύψουμε μέσω του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να γνωρίζω είναι αν μπορούμε να έχουμε και μια ποιοτική ανάλυση όσον αφορά τις κρίσεις εκείνες τις οποίες δεν καταφέραμε παρκώς να καλύψουμε διότι δεν είχαμε τα παρέτα κονδύλια. Το είπα και πριν από λίγο στα πλαίσια της συζήτησης για τη γνωμοδότηση του κυρίου Λίτς και θα έχω και άλλα πράγματα να πω στο μέλλον όσον αφορά την στάση του Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε περήφανοι. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά πολιτικά να επικρίνουμε το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενσωματώσει τη στάση του Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να επικρίνουμε αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο, το οποίο πραγματικά δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο ύψος των περιστάσεων. Το λόγο είχε ο κύριο Λίτ και στη συνέχεια θα απαντήσει ο κύριο Φερνάντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε κύριε Φερνάντε. Ε, είμαι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση να τοποθετηθώ σύντομα. Θέλω να προβάλλω ένα θέμα, δηλαδή ε, το όλο και μεγαλύτερο κενό ανάμεσα στις υποχρώσεις ε, και τις ε, πληρωμές. Αυτά τα οποία μας είπατε σχετικά με την χρηματοδότηση που δεν καταβάλλεται, παραδείγματος χάρη για την επισητιστική βοήθεια, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και έχοντας κατά νου ότι φέτος είναι η χρονιά της ανάπτυξης και έχουμε φτάσει ε, ήδη κατά το πρώτο εξάμεινο σχεδόν στο ανώτατο όριο της χρηματοδότησης ε, που μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα δηλαδή τίθεται το θέμα ε, κυρίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό που είπε και ο κύριος Νόζα, το πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρηματοδότηση. Κύριε Φερνάντες, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημεριζόμαστε τους στόχους στους οποίους αναφερθήκατε όσον αφορά τώρα το ρόλο του Συμβουλίου και το ρόλο μεμονωμένων κρατών μελών. Γνωρίζετε ότι εγκρίνουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται ομοφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου. Πρέπει να συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε στη συνέχεια ένα προπολογισμό όμως, ο οποίος είναι πολύ πιο μικρός από αυτό που προβλέπεται στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου σε αιτήσια βάση πώς είναι ποτέ δυνατόν τα κράτη-μέλη τα οποία ομόφωνα ενέκριναν συγκεκριμένο όριο επίπεδο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίνουν στη συνέχεια ετήσιο προπολογισμό ο οποίος υστερεί, ο οποίος υπολείπεται του ποσού που έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κατονομάσουμε τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη που συνεχώς και συστηματικά στρέφονται κατά του ετήσιου προπολογισμού της Ένωσης. Στα πλαίσια τώρα τη ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε έναν ξεχωριστό προπολογισμό και έχουμε βέβαια και τον εθνικό προπολογισμό των κρατών μελών. Γιατί ξέρετε ότι και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα ακολουθούν πολιτική, εθνική όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία από μόνα τους μειώνουν τη δική τους επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό αποτελεί εθνική τους αρμοδιότητα και εθνική τους ευθύνη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των πληρωμών, το 2014 είχαμε 650 εκατομμύρια ευρώ καθυστερούμενες πληρωμές. Πραγματικό όνειδος είναι αυτό, αναφέρομαι στο τμήμα 4. 650 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν είχαν εξοφληθεί, δεν είχαν καταβληθεί. Πραγματικό όνειδος είναι αυτό. Καταλαβαίνετε ότι διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία μας. Η αναλήψη υποχρεώσεων θα πρέπει να παίρνει τη μορφή πληρωμών στη συνέχεια. Αυτό αποτελεί υποχρέωση δική μας, νομική μας υποχρέωση και δέσμευση. Έχουμε επιμείνει πάρα πολύ στο ζήτημα των πληρωμών. Ξέρετε ότι έχουμε μια διοργανική συμφωνία με το Συμβούλιο ακριβώς για το ζήτημα αυτό της ουσιαστικής καταβολής των πληρωμών. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι οι διοργανικές αυτές συμφωνίες, οι οποίες είναι εγγραφές, ελπίζω ότι τουλάχιστον μη τι άλλο αυτές οι συμφωνίες θα τηρούνται από το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει τεράστιες μάχες ε, για τις πληρωμές αυτές και για το περιθώριο έκτακτης ανάγκης και απαιτούμε όλο και πιο ισορροπημένους προπολογισμούς, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι το Συμβούλιο επιμένει σε περικοπές, τις οποίες δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δείτε στο τμήμα 4, τη γραμμή 21.02.04.05, μετανάστευση και άσυλο, βλέπετε ότι στις πληρωμές έχουμε μία περικοπή της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ανάληψη υποχρεώσεων είναι 200 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε εδώ πέρα τι γίνεται, τη στιγμή που το Συμβούλιο αυθαίρετα τελικά παίρνει κάποιες γραμμές του προπολογισμού και λέει ότι εδώ πέρα θα κάνω περικοπές ή σε κάποιες άλλες γραμμές του προπολογισμού δεν θα κάνω περικοπή για να στείλω ένα θετικό πολιτικό μήνυμα. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένε τροπολογίες, προφανώς θα συμπεριληφθεί και η δική σας εγγνωμοδότηση στην εντολή που μου δίνετε και προφανώς θα εξετάσουμε τη συμβολή της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια του προπολογισμού και στα πλαίσια των προκλήσεων που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Θα πρέπει βέβαια να εξετάσουμε και τις τροπολογίες όλων των επιτροπών και της δικής σας βέβαια της Επιτροπής. Έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο στη διαθεσή μας, θα πρέπει να παραμείνουμε σε συνεχή επαφή. Και βέβαια, αφού κατατεθούν οι τροπολογίες και αφού περάσουμε και στις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου πάντα το στόχο της εξωτερικής αλληλεγγύης. Η εξωτερική αυτή αλληλεγγύη αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της εντολής μας, η ανθρωπιστική αναπτυξιακή βοήθεια είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να δεχθούμε εκτόσεις στον στόχο αυτό, σε όλα αυτά δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Κύριε Γκέρενς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι δεν μπορέσαμε να επιτελέσουμε ακριβώς επειδή δεν είχαμε τους απαραίτητους πόρους. Και αυτό συνάδει με αυτά που είπα πριν από λίγο. Όταν δεν πράττουμε κάτι και όταν παραλείπουμε να το κάνουμε συστηματικά, τότε το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αν είχαμε όντως αναλάβει δράση καταβάλουμε ένα πολύ σημαντικό τίμημα για την απραξία, για την απουσία δράσης και πολλές φορές το τίμημα αυτό, το τίμημα αυτό είναι πολύ ψηλότερο από το πραγματικό κόστος της δράσης αυτής. Για παράδειγμα, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα παιδείας. Έχουμε φτάσει στον απίστευτο αριθμό των 4 εκατομμυρίων παιδιών από τη Συρία που έχουν χάσει τα πάντα βέβαια αν εμείς μείνουμε άπραγοι, καταλαβαίνετε ότι το τίμα που θα καταβάλουμε στο μέλλον, το μέλλον θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Ανταυτού πρέπει αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουμε μια δράση για αυτό τον τομέα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έχοντας ως στόχο να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προπολογισμό και να έχουμε ένα προπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τις υποχρεώσεις μας, θα τηρεί τους κανόνες, θα τηρεί τις δηλώσεις που κάνει το Συμβούλιο, που θα τηρεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, που θα τηρεί και θα σέβεται όλα τα μέσα ευελιξίας που υπάρχουν, καθώς επίσης και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της εντολής μας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον στόχο αυτό της εξωτερικής ελληνική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Φερνάντε, Από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε όλοι με αυτά τα οποία είπατε. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της συζήτησής μας για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και να δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στον κύριο Λίτς. Ευχαριστώ. Να πατήσω στα τελευταία σημεία. Θα τα πω όμως στα γερμανικά, γιατί είναι πιο εύκολο για μένα και θα βασιστώ και στα θέματα της εκπαίδευσης γιατί είναι προτεραιότητα και για μας ε, και, αυτό το θέμα για εμάς. Συνεχίζω λοιπόν στα γερμανικά. Thank you to all colleagues to have contributed uh, until this point. Uh, in... Uh, λοιπόν, ε, πριν περάσω στις ε, τροπολογίες του προϋπολογισμού θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο βασικά προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν και αυτά θα πρέπει να έχουμε κατά νου στις ε, τροπολογίες. Στις συζητήσεις και στις ε, τριμερείς συζητήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα προβλήματα. Το πρώτο που είπα είναι το ε, διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να το αντιμετωπίσουμε περισσότερο το 2016. Αν λοιπόν οι πληρωμές παραμένουν μικρότερες από τις υποχρεώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερής πληρωμών, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε όλοι. Άρα δηλαδή και καθυστέρηση προγραμμάτων. Ε, το βρίσκω πολύ σωστό, να προσπαθήσουμε να το φύγουμε αυτό ε, και να ε, κάνουμε και μελέτες αντικτύπου αν προκύπτει προκύψουν ε, καθυστερήσεις. Σας είπα, οι περικοπές μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις πληρωμών. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε τις ε, προτάσεις του Συμβουλίου προς την Επιτροπή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι οι ε, αυξανόμενε συγκρούσεις, ε, στο Ιράκ, ε, στο Σουδάν και θα έχουμε περισσότερους πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφική κατάσταση και να αυξήσει τα κονδύλια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Συμβούλιο λειτουργήσε σωστά και δεν έκανε περικοπές. Ε, ως εισηγητής βέβαια εγώ ε, θα ζητήσω αύξηση του προπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια και η τροπολογή μου είναι η εξή. Ζητώ στα περισσότερα εργαλεία TCI ε, να επανέλθει ο προπλογισμό σε αυτά που πρότεινε η Κομισιόν. Ε, σε τρία συγκεκριμένα εργαλεία προτείνω αύξηση του προπλογισμού και όπως αναφέρθηκε αυτά είναι το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου. Εκεί ο προπολογισμό πρέπει να αυξηθεί ε, ξεκινώντας από την πρόταση των Κομισιών ε, σε 45 εκατομμύρια και 250.000 ε, στις υποχρεώσεις και 22 εκατομμύρια και 560.000 στις πληρωμές. Να πάμε στα 49 εκατομμύρια και 775.000 υποχρεώσεις και 25 εκατομμύρια και 60.000 στις πληρωμές. Αυτές να είναι οι αυξήσεις. Οι τοπικές αρχές ξεκινώντας από την πρόταση Κομισιόν των 60 εκατομμυρίων, 291 εκατομμύρια στις υποχρώσεις και 18 εκατομμύρια στις πληρωμές κατά την δική μου την τροπολογία να πάμε στα 66 εκατομμύρια και 291.000 στις υποχρώσεις και 20 εκατομμύρια και 116.000 στις πληρωμές. Ο λόγος είναι ότι ε, μετά το 2015 θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και οι τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν κατά το μέγιστο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται εκπαίδευση και κατά τη διαφθορά σε βελτιωμένη υποδομή έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η τρίτη τροπολογία αφορά την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις στις περιοχές σύραξης είναι τεραστίων διαστάσεων. Στο Ιράκ έχουμε 8 εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. 55 εκατομμύρια ευρώ, άρα δηλαδή ο προϋπολογισμός αυτός πρέπει να διαθέσει ταχύτατα πόσιμο νερό, φάρμακα, είδη υγιεινής, δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων και ένα άλλο κομμάτι στην εκπαίδευση όπως αναφέρθηκε ήδη από διάφορους ομιλητές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1,95% της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εκπαίδευση. Αυτό το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί. Οι σοσιαλδημοκράτες απαιτούν τα 10 εκατομμύρια των 55 εκατομμυρίων να διοχετευτούν στην εκπαίδευση. Άρα δηλαδή κινητά σχολεία και ε, δυνατότητα τα παιδιά και στη Συρία να μπορούν να πηγαίνουν ε, παρόλα αυτά στο σχολείο για να εκπαιδευτούν. Αυτά όσον αφορά τα κεντρικά θέματα που θέλω να προβάλλω. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους Επιτροπής και την Επιτροπή Προεπολογισμού για τη συνεργασία και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και περαιτέρω. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα που αναφέρθηκαν χτες, ε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ε, ποια προγράμματα μπορούν να παραταθούν το 2016 αυτού θα τοποθετηθώ σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί έτσι ώστε η γνωμοδότηση να έχει φτάσει σε εσά πριν από την διορία κατάθεσης τροπολογιών που είναι η 27η. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τους κοιόδης. Ο κύριος Γκέρενς καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διστάζω πώς να το χαρακτηρίσω, ε, λίγο καθησυχαστικό, ανησυχητικό το σχέδιο αυτό προϋπολογισμού. Δεν σέβεται τις δεσμεύσεις στο Συμβούλιο. Και μας λέει παραμύθια. Σας υπενθυμίζω. Τι μας είπε για το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο. Δεν πήραμε στο 4 αυτό που θέλαμε. Ο Βον Ρομπάι ήρθε στη διάσκεψη των Προέδρων που ήταν ανοιχτή για όλους τους βουλευτές και μας είπε ναι παραδέχομαι ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά σας. Τα κράτη-μέλη όμως αποζημιώθηκαν με βάση κάποια χρήματα και κάποιες δεσμεύσεις για, το, για την περίοδο αυτή. Όμως τη βλέπουμε κατά μέσο όρο των ε, εισφορών. Εδώ έχουμε μείωση. Άρα μας λένε παραμύθια. Τι σημαίνει, τι γίνεται επί της ουσίας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει η Ευρώπη. Αν βγείτε και πάτε στην πλατεία του Λουξεμβούρου έξω από το κοινοβούλιο, ο πρώτος που θα σας πει τι κάνουμε για να τα σε δυνητικές κρίσεις του χρόνου, θα πούμε δεν έχουμε αρκετά χρήματα στον προπολογισμό. Και γι' αυτό θα κατηγορηθεί και θα στιγματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπατε και εσεί, κύριε Φερνάντε, στην εισαγωγική σα ομιλία, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να στιγματίσουμε. Αυτά φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία. Αυτά φέρουν την ευθύνη γιατί δεν μπορούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Μπορεί να λέμε μεγάλα λόγια για τις προτεραιότητες, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η μόνη λύση αν θέλουμε πραγματικά να αποκριθούμε στα αιτήματα που θα έχουμε και του χρόνου. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε όλους τους πόρους που έχουν εγγραφεί στον ε, προπολογισμό του χρόνου για να τα αποκριθούμε στις κρίσεις και όχι για να απορροφήσουμε με το προηγούμενο ετών. Όλοι ε, θέλουν νέα στρατηγική για τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά τα πράγματα, να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μα γίνεται αυτά να τα πετύχουμε με λιγότερα χρήματα. Που πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα αν δεν δίνουμε τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν τα κράτη-μέλη αρνούνται να συμμετάσχουν και το βλέπουμε. Με το που ξεκινάει η συζήτηση για την αλληλεγγύη, για τους καταβλισμούς προσφύγων, βλέπουμε πώς ε, διχάζονται τα κράτη-μέλη. Επίσης, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, όταν τεθούν σε ισχύ, θα έχουμε απομείωση της αξίας, ε, ιδίως για τα αφρικανικά κράτη. Άπαξ και τεθούν σε εφαρμογή και επικυρωθούν οι συμφωνίες αυτές, θα έχουν σε αποτέλεσμα λιγότερα έσοδα για τις χώρες εταίρους. Μπορεί να λέμε ότι από το ΕΤΑ μπορούμε να τις σταθμίσουμε τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου της απόλυσης, είτε τη σχετικό κονδύλιο. Και είναι αλήθεια αυτό. Όμως το κονδύλιο αυτό άπαξ και εκταμιευτεί για να τις σταθμίσει τις απόλυες των χωρών, θα λείψει ε, το ποσό αυτό από άλλα κονδύλια. Ξέρουμε πόσο απαραίτητο είναι στι λιγότερο προηγμένες χώρες κυρίω να βελτιώσουμε το σύστημα υγεία. Από πού θα έρθουν τα χρήματα λοιπόν. Και μπορώ να πω και πολλά άλλα. Άρα, συμπέρασμα. Α πάψουν να μας λένε παραμύθια και α ασκήσουμε κι εμείς ε, κριτική, ε, όχι με αγενή τρόπο, αλλά ας είμαστε πάντως ε, ομοί. Να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να τα πούμε χήμα. Και έχουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Εκεί πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις μας, διότι προσπαθεί να μας ε, ε, ρίξει στάχτη στα μάτια με ό,τι μας λέει το Συμβούλιο, που λέει άλλα αντί άλλων. Μας λέει δεν είχατε αρκετά στο CFP, θα το πάρετε γιατί θα έχουν ε, περισσότερη συμμετοχή τα κράτη-μέλη. Ε, όλα αυτά είναι κοροϊδία. Okay, thank you and... Uh, <coughs> Σας ευχαριστούμε κυρία Χάουτα, αλλά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες αυξήθηκαν στις γραμμές του προπολογισμού που έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό μας διευκολύνει να καλύψουμε τις καθυστερούμενες πληρωμές και τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Επίσης, έχουμε 261 εκατομμύρια ευρώ στο EFF στο τμήμα 4 του προπολογισμού και γι' αυτά προβλέπεται ένας βαθμός ευελιξίας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο κάποιους στόχους ε, τους οποίους όμως θα πρέπει να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά. Ας έχουμε επίσης κατά νου ότι και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θέλει και αυτή να αυξηθούν οι πιστώσεις ε, στον προπολογισμό που έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή βοήθεια. Ιδίως όσον αφορά την ε, Παλαιστίνη. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα δούμε κάποιες ε, αυξήσεις. Αυτό ελπίζω τουλάχιστον. Επίση, είναι θετική η εξέλιξη το ότι έχουμε περισσότερες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να πάνε προς τις τοπικές αρχές όπως πρότεινε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμως προκαλεί μια κάποια ανησυχία είναι ότι στα πλαίσια του μέσου ανεπτυξιακής βοήθειας υπάρχουν μειώσεις όσον αφορά τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και όσον αφορά τις πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι πιστεύω προβληματικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, όσον αφορά τις ε, διοικητικές δαπάνες και τις σχετικές πιστώσεις, ξέρετε ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και για αυτές τις δυτικέ δαπάνες. Εδώ πέρα έχουμε μία αύξηση και θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό. Τώρα, για τις χώρες εκείνες όπου το μέσο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις χώρες της Νοτιού Αμερικής, οι οποίες δεν αποτελούν αυτή τη στιγμή χώρες προτεραιότητας όσον αφορά την πολιτική ενεπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μιλήσαμε πολύ για την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επενδύσει περισσότερο στη Συρία και ιδίω να βοηθήσει τα παιδιά της χώρας αυτής και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μία εντελώς χαμένη γενιά σε αυτή τη χώρα. Αναφέρομαι στα παιδιά εκείνα τα οποία δεν θα καταφέρουν ποτέ να πάνε σχολείο και να εξελιχθούν ως ενήλικες. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε όλα τα κονδύλια που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη χώρα αυτή. Ο κύριος Φερνάντες αλλά και ο κύριος Λίτς αναφέρθηκαν στο ζήτημα της μετανάστευσης και για τον τομέα αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες πιστώσεις. Πρόεδρος. Κυρία Χόιμπερ, παρακαλώ. Θέλω να δείξω και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε και αναφέρθηκε και προηγουμένως ε, ότι υπάρχει μια ε, γραμμή σχετικά με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυξήθηκαν εκεί τα κονδύλια. Από την άλλη όμως περιορίζουν τα κονδύλια ε, σχετικά με την προστασία του κλίματος. Ε, αυτό θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα που θα είναι το θέμα του μέλλοντος και θα χαιρόμουν πάρα πολύ εάν μπορούσαμε για αυτό το θέμα να αφήσουμε τα κονδύλια ως έχουν. Πολύ ωραία. Ε, δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο, τουλάχιστον όχι στον καταλογό μου. Ο κύριος Λίτς θα ανακεφαλαίωσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ε, πιστεύω ακριβώς αυτό που είπατε Δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε στο πώς ακριβώς επιθυμούμε να συνεχιστεί η κατάσταση στα οικονομικά, ε, να δούμε τι προσπάθειες ε, πρέπει να καταβάλουν οι Ευρωπαίοι. Επίσης αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μας ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό ε, πράγματι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των ε, προεπλογισμών. Όσον αφορά την έκθεση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας για το τι μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε στον προεπλογισμό της επόμενης χρονιάς και προσβλέπω στο να συζητήσουμε στο μέλλον για το κλίμα να το δούμε και αυτό λιγάκι έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω μήπως επιθυμούν ε, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να σχολιάσουν κάτι. Παρακαλώ. Ε, δεν έχουμε ερωτήσεις να κάνουμε. Θέλουμε μόνο να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας ε, για το ότι θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες, θα αυξηθεί περαιτέρω ο προϋπολογισμός, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς τις προτεραιότητες ε, για την επόμενη χρονιά. Γνωρίζετε ότι κατά κανόνα το 20% ε, παρακρατείται σε ένα ειδικό απόθεμα ήδη από την αρχή της χρονιάς ε, για να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει νέες κρίσεις. Βέβαια υπάρχει και το απόθεμα έκτακτων αναγκών. Αυτό είναι για μεγαλύτερης ε, κρίσης την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν προβλήματα γιατί υπάρχουν ήδη υποχρεώσει που απορρέουν από το παρελθόν κυρίως σε σχέση με τη Συρία και τη στρατηγική της Επιτροπής που παρουσιάστηκε σε αρχές του έτους. 1,1 δις θα προσθεθούν και άλλα. Και επίσης έχουμε και άλλα 100 εκατομμύρια από τα 900 τόσα ε, Άρα δηλαδή μιλάμε ότι θα υπάρξει θέμα χρηματοδότησης. Εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε να αυξήσουμε περαιτέρω κυρίως ε, τη νέα προτεραιότητα για την εκπαίδευση σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια, οποιαδήποτε τέτοια βοήθεια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που κατευθύνουν τα χρήματα και κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση έχουμε κάνει πολύ καλή εμπειρία ε, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά και την ε, πρωτοβουλία ειρήνης. Υπάρχουν νέες παρεμβάσεις ε, στο θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης και της παιδείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, πρωτοβουλίες σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, οπουδήποτε κριθεί αυτό απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι. θα πάρετε το σχέδιο γνωμοδότησης και προθεσμία για να το τροποποιήσετε θα έχετε έως την 1η Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Οι δημοσιονομικές τροπολογίες θα ψηφιστούν στις 3 Σεπτεμβρίου την ίδια ημέρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τη γνωμοδότηση. Αυτά είναι αυτές οι ημερομηνίε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε 10 λεπτά για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία γιατί προβλεπόταν να αρχίσει 11 και 4 η ψηφοφορία. 10 λεπτά διάλειμμα.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 Uh, ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Προτού όμως το κάνουμε αυτό, ας ελέγξουμε αν λειτουργούν καλά οι συσκευέ μας. Και μετά την ψηφοφορία συνεχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Όσοι συμφωνείτε λοιπόν με αυτό μπορείτε να ψηφίσετε υπέρ, όσοι διαφωνείτε μπορείτε να ψηφίσετε κατά. Και ψηφίζουμε και έτσι δοκιμάζουμε τις συσκευές. Άρχιτη ψηφοφορία. Ο κύριος Πρέντερ δεν έχει την κάρτα του μαζί του. Λοιπόν, έχουμε μόνο μία ονομαστική κλίση στο τέλος, αλλά λειτουργούν από ό,τι βλέπω συσκευέ συσκευές. Πέρας. Κανιά υπέρ, ουδής κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ρόλο των τοπικών αρχών στι αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Η κυρία Ελένη Θεοχάρου είναι η συγγήτρια. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 9. Διορθώνει ο Πρόεδρος, τροπολογία 27, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Διορθώνει ο Πρόεδρος, τροπολογία 28, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 έχει αποσυρθεί. η 38 λοιπόν υπέρ, κατά,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 Πολλές αποχές βλέπω. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την τροπολογία 44. Άρτη ψηφοφορία. Κρίνεται. 12 υπέρ και 2 κατά 9 αποχές. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ορισμένοι ψήφισαν μάλιστα και δύο φορές. γιατί 45 ψηφίσαμε υπέρ πάλι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Αυτή έχει αποσυρθεί. Περνάμε λοιπόν στη 47 υπέρ. 47 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει. Άρα περνάμε στην τροπολογία 67. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Περνάμε στην αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16, 17 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 άρθρη ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε τώρα στις θεολογικές αναφορές 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα για το σύνολο του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόκειται για νομαστική ψηφοφορία, άρχτη ψηφοφορία. Πέρας, 19 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες κατά αυτόν τον τρόπο και όπως συμφωνήσαμε συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα φύλλο και ανάπτυξη. Συγχαρητήρια, στη, συγχαρητήρια στην κυρία Θεοχάρους. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, φύλλο και ανάπτυξη. Εδώ έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προφορική ερώτηση και ψήφισμα για την περάτωση της συζήτησης όσον αφορά το ζήτημα αυτό σχέση μεταξύ της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης. Θα θυμάστε ότι με εξωτερικούς ομιλητές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίασή μας και οι συντονιστές είχαν πει ότι στη συνεδρίαση της 23ης ε, Ιουνίου θα παρουσίαζαν προφορική ερώτηση καθώς επίσης και ψήφισμα για την περάτωση της συζήτησης. Και ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο δράσης όσον αφορά το φύλλο και την ανάπτυξη για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μπορείτε να δείτε τις δύο αυτές προφορικές ερωτήσεις, η μία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η άλλη απευθύνεται στο Συμβούλιο. Τις έχετε και τις δύο στους φακέλους σας και βλέπετε ότι και οι δύο προφορικές ερωτήσεις αλλά και το σχετικό ψήφισμα αναφέρονται σε κάποιες αδυναμίες και προβλήματα που υπάρχουν στο εφιστάμενο σχέδιο δράσης και ζητούν ανανεωμένη πολιτική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το νέο σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια όσον αφορά το ζήτημα των της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης. Να δώσω καταρχάς το λόγο στην συγκήτριά μας για το gender mainstreaming στην κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Λίντα Μακάβαν, η πρόεδρος μας, είναι στην Αντίσα Μπέμπα, κεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τη χρηματοδότηση, για την ανάπτυξη, για τη διάσκεψη που γίνεται εκεί. Προετοιμάσαμε από κοινού το σχέδιο ψηφίσματος ε, και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης για το φύλλο είναι μια πολύ ε, σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να απολέσουμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διάσταση του φίλου ως ένα εγκάρσιο ζήτημα και ειδικό θέμα και για την πολιτική της συνεργασία για την ανάπτυξη. Και ιδίως σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο αντιπροσωπείας. Ε, νομίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις από την κοινότητα των πολιτών μέχρι και την αξιολόγηση της Κομισιόν ε, για το σχέδιο δράσης ε, συμφωνούν ότι θέματα δεν λείπουν. Ε, πολλά καλά θεματικά ζητήματα έχουμε για την οικονομική από την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μέχρι τα δικαιώματα των γυναικών για τη σεξουαλική αναπαραγωγική τους και το καθεξής. Αυτό που λείπει είναι οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη. Και αυτός είναι και ο τόνος της πρώτης ψηφίσματος. Γιατί θέλουμε, θέλουμε να κατεθεί το Σεπτέμβριο, όπως και μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα αξιολόγηση του τρέχοντος σχέδιου δράσης ε, για το φύλλο. Νομίζω ότι είναι η Κομισιόν ε, διατεθειμένη να σημειώσει και να διδαχθεί από, τα μέχρι τώρα, ε, από τις εμπειρίες. Και το βασικό μάθημα είναι ότι δεν ε, έχουμε φέρει σε πέρα στις δεσμεύσεις μας. Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεσμεύσεων και της δυνατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει αποτελέσματα. Επίσης οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η ηγεσία της ΕΙΕΔ και της δίκησης δεν έχουν καταφέρει να μεταδώσουν επικοινωνιακά τις προτεραιότητες ούτε στο προσωπικό ε, της έδρας ε, των κεντρικών ούτε στις αντιπροσωπείες. Άρα δεν καταλαβαίνει το προσωπικό τι σημαίνει στην πράξη πολιτική για το φύλλο και νομίζω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα διορθώσουμε αυτά. Ζητούμε μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην το πάρει ελαφρά το όλο θέμα. Αλλά το κοινοβόλιο πρέπει να ζητήσει να υπάρξει ανακοίνωση. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Επίτροπος Μιμίτσα, ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Ανάπτυξη, δεν θα ήταν καθόλου αντίθετος σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν, θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να αποδώσουν τη δέωσα προσοχή στο πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό της πολιτικής Συνεργασία για την ανάπτυξη. Αν θέλουμε λοιπόν καλύτερη νομοθεσία, πρέπει να πιέσουμε, να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν που φαίνεται να διστάζει και πρέπει να την ε, ενθαρρύνουμε να προβεί σε αυτή την ανακοίνωση, διότι με την ε, ε, αναντιστοιχεία δεσμεύσεων και δράσεων πλέον είναι καιρός να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και τώρα ε, καταρχήν θα λάβουν το λόγο οι σκιώδεις συγητές. Όχι, οι συντονιστές, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Και ξεκινάμε με τον κύριο Charles Γκέρενς. Ο Charles παρακαλώ. Δύο πράγματα μπορώ να πω. Πρώτον, ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος Χάιντι. Και δεύτερον, δεν είμαι σκιώδης για το θέμα αυτό. Μόλις και διάβασα τα σχετικά, αλλά με πείθει η Χάιντι με αυτά που είπε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Οι άλλοι συντονιστές ο κύριος Ντέβα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλάμε για κάτι το οποίο θίγει πολλά και ενδιαφέροντα. Μιλάμε δηλαδή για κάτι ε, το οποίο είναι προφανές. Ε, το θέμα του φύλου, κυρίως ο ρόλος των γυναικών ε, στην ανάπτυξη, είναι καθοριστική σημασίας σε όλες τις κοινωνίες, στην Αφρική, ο ρόλος της γυναίκας ε, στην οικογένεια, ο ρόλος της ε, γυναίκας στην ανατροφή των παιδιών, στην ε, μετάδοση αξιών, καλή συμπεριφοράς, αστικής υπευθυνότητα, ο ρόλος τους είναι πραγματικά καθοριστική σημασίας. Κυρίως ο ρόλος των γυναικών στην Αφρική ε, που κερδίζουν ε, και χρήματα για την οικογένεια. Στην Κάνα, στην Ανατολική Αφρική, οι γυναίκες είναι εκείνες ε, που διαχειρίζονται τις μικρές επιχειρήσεις και την οικονομία και άντρες κάθονται στο καφενείο και τα λένε και δεν φέρνουν λεφτά στο σπίτι. Εδώ μιλάμε για θέμα νοτροπίας ε, και ο ρόλος των γυναικών κυρίως στην Αφρική και σε κάποιον τρόπο και στην Ανατολική Ασία είναι καθοριστική σε σημασία. Αν πάτε ας πούμε σε εργοτάξιο στην Ινδία θα δείτε τις γυναίκες ε, να κουβαλάνε τα ε, τούβλα και οι άντρες δεν κάνουν τίποτα, κάθονται, ξεκουράζονται, λιάζονται. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση. Οι άνδρες ε, να μην είναι πια τεμπέληδες, ε, να αναδιοργανωθούν αν θέλουν να συμμετέχουν ε, στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Και έχω συναντήσει πολλές περιπτώσεις στη Σρι Λάνκα, όπου οι άνδρες από τα 20, συγγνώμη, ναι, από τα 20 μέχρι τα 40 δουλεύουν και μετά λένε ότι στις γυναίκες ότι πάνε στην, ε, σε χώρες, στο σπίτι κάποιου έχει για να δουλέψει εκεί και μετά συνταξιδετούνται. Η γυναίκα λοιπόν εκείνη που κρατάει την οικογένεια ε, και ο τύπος κάθεται σπίτι του. Αυτή λοιπόν η τροπία πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να ε, μετατεθούν οι ευθύνε στον άντρα, ο άνδρας να έχει τις ίδιες ευθύνε ε, όπως και οι γυναίκες ε, σε αυτούς τους πολιτισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ίσως αυτό να φαίνεται στον υπεριαλισμό ή οπουδήποτε αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αν οι άνδρες και οι γυναίκες είναι πραγματικά ίσοι, δηλαδή οι γυναίκες να μην τρομοκρατούνται στο να αναλαμβάνουν όλες αυτές τις ευθύνες γιατί τους λένε να πάνε στη Μέση Ανατολή ε, τους λένε να κουβαλάνε τα τούβλα και όλα τα άλλα τα φρικιαστικά ε, όπου ο άνδρας ε, λέει τι πρέπει να κάνει η γυναίκα, αν της πει η κουβάλα σαν το σύσυφο τα τούβλα μέχρι την κορυφή του βουνού και ξανακατέβα, θα το κάνει. Αυτό είναι λάθος λοιπόν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες. Αυτή όλη η δομή είναι παντελώς άδικη και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέμα δεν είναι να μιλάει κανείς με τις ε, κεντρικές κυβερνήσεις. Αυτές είναι πολύ μακριά από το πρόβλημα. Ε, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή συνομιλούμε με τις κεντρικές κυβερνήσεις που είναι πολύ μακριά από το πρόβλημα, ενώ κατ' ουσίαν αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί επί πρέπει να έρθουμε σε επαφή με δήμους και κοινότητες ε, που διαχειρίζονται τα χωριά και από αυτούς να περιμένουμε, σε αυτούς να εκφράσουμε τις προσδοκίες μας. Αυτές οι φλιαρίες ε, με τις ε, κεντρικές κυβερνήσεις δεν οδηγούν πουθενά και κανένας κανένας ε, υπουργό, κανένας κυβερνητικός δεν θα πάει σε ένα χωριό να πει στις γυναίκες ε, σταματήστε να κουβαλάτε τα τούβλα. Μιλάμε λοιπόν ε, στις κεντρικές κυβερνήσεις και δεν αλλάζει τίποτα. Αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να δουλέψουμε σε επίπεδο βάσης, με τις τοπικές ΜΚΟ, με τις ε, τοπικές κοινωνίες των πολιτών και να επιδιώξουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη βάση της. Ο συντονιστής της Γκουε μόλις βγήκε έξω. Η Μαρία Φόιχουφ εκ μέρους των Πρεσίνων είναι η επόμενη. Εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ισότητας των δύο φίλων. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ε, έκθεση που εκπονήθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια μετά από εντολή των ΗΠΑ για το θέμα, για τον τομέα της γεωργίας. Και εκεί τέθη η διάσταση του φίλου και καταλήξαν στο ότι αν ένα δολάριο το δώσει κανείς σε έναν άντρα είναι πιθανό να χαθεί το δολάριο. Αν το δολάριο το δώσει κανείς σε μια γυναίκα θα λάβει πίσω 3 δολάρια. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες στις οικονομίες των κρατών. Δεν πρέπει βέβαια να γνωρούμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες ε, όπου στις γυναίκες δεν επιτρέπεται να είναι γεωκτήμονες γενικά να κατέχουν ιδιοκτησία. Είναι και θέματα πολιτιστικά, είναι θέματα πολύ σημαντικά ε, κυρίως όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της φτώχειας, πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ενέργειές μας και τις γυναίκες. Και όλα θα λειτουργήσουν μόνο αν οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας είτε στην παραγωγή είτε οπουδήποτε αλλού. Πρόκειται για ένα πολύ βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της φτώχειας, της ε, ανόρθωσης οικονομιών. Ε, γι' αυτό λοιπόν υπογραμμίζω για άλλη μια φορά ε, το πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση και ευελπιστώ να έχουμε και αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται όμως πάρα πολλοί συνάδελφοι για το ζήτημα αυτό. Τρεις μόνον συντονιστές που έχουμε εδώ πέρα. Κανείς από τους αριστές, κανείς από το ΕΛΚΑ, άλλοι πάλι απουσιάζουν. Υπάρχει κάποιος άλλος πάντως που θα ήθελε να πάρει τώρα το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως. Πείτε μας ποιος είστε, παρακαλώ πολύ. Ε, από την DG Justice από την ε, Μονάδα για την Ισότητα, ίσως από την ΤΕΦΚΟ όμως θα ήταν καλύτερα να σας μιλήσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ε, ζητώ συγγνώμη. Ξεκίνησε νομίζω λίγο νωρίτερα η συνεδρίαση αυτή από ό,τι περιμέναμε. Δεν έχει φτάσει ακόμα ο αρμόδιος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περίμενε ότι θα το καλύπτεται λίγο αργότερα αυτό το σημείο. Κανένα πρόβλημα τότε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χάουταλα. Δύο παρατηρήσεις. Ο κύριος Ντέβα έχει απόλυτο δίκιο όταν περιγράφει κατά αυτόν τον τρόπο την κατάσταση των γυναικών στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα όμως να απαντήσω και λίγο στις δικές σας παρατηρήσεις όσον αφορά τους μεμονωμένους αυτούς δράστες και το γεγονός ότι θα πρέπει όντως να έρθουμε σε επαφή με τις επαρχιακές τοπικές κυβερνήσεις. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουμε ότι ε, τα συντάγματα των χωρών αυτών ιδιαίτερα προδευτικά όσον αφορά την ισότητα των ε, ανδρών και των γυναικών. Για παράδειγμα προβλέπεται ένα ελάχιστο έτος, μια ελάχιστη ηλικία όσον αφορά τον γάμο τα 18 έτη. Αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη, στο εφιστάμενο δηλαδή δικαστικό σύστημα παρακάμπτεται ο νόμος αυτός και έχουμε βέβαια το πρόβλημα αυτό των γάμων των παιδιών που θεωρώ ότι αποτελεί πραγματικά καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Έχετε λοιπόν δίκιο. Είδα επίσης ότι στο Μαλάουι υπήρχε ένας ε, ηγέτης τοπικός, από τον οποίο ζητήθηκε να παντρέψει πολλά νεαρά κορίτσια, τα οποία προφανώς ήταν κάτω των 18 ετών, και αποφάσισε να τα στείλει όλα στα σχολεία ανταυτού και είπε ότι κοιτάξτε έχουμε ένα σύνταγμα, πρέπει να αλλάξουμε πλέον τις πρακτικές που ακολουθούμε, δεν είμαστε πλέον μια χώρα στην οποία τα νεαρά κορίτσια απλώς τα παντρεύονται πιο ηλικιωμένους άνδρες και θα σταματούν να πηγαίνουν στο σχολείο και θα ασχολούνται μόνο με τα οικιακά. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε κάποια θετικά παραδείγματα επιτόπου τα οποία θα πρέπει προφανώς να χαιρετήσουμε και να ενθαρρύνουμε. Και θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να μιλούσα με την γυναίκα αυτή ηγέτη μιας κοινότητος στο Μαλάουι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να θαρρύνουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή στρέφονται κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο όνομα της παράδοσης, στο όνομα των εθήμων. Είμαι συντηρητική αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να ταχθώ υπέρ του γάμου όταν ο γάμος αφορά ανήλικα κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πολύ Χάιντι, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 2η Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Η προφορική ερώτηση θα ψηφιστεί στις 22 Σεπτεμβρίου και το ψήφισμα προφανώς. Ολοκληρώνεται τώρα η συνεδρίασή μας και θα συνεχίσουμε πάλι στις 3 το μεσημέρι. Λύεται η συνεδρίαση.